θέλω να σας τη διαβάσω. Δηλαδή οι αρμόδιες αρχές της Ιρλανδίας ανακοίνωσαν ότι ο κύριος Σίας Ντερόσα από τις 15 ε, Φεβρουαρίου του 2012 ε, θα αντικατσαθεί από την κυρία Κοστέλο και εγώ ε, καλωσορίζω την ναι, έρχονται, δεν ξέρω ήρθε ήδη εδώ είναι γεια σας χαίρετε καλώς ήρθατε Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού του Κοινοβουλίου όλα τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδρίες του Κοινοβουλίου με πλήρη δικαιώματα όσο η ε, θητεία τους ε, δεν αμφισβητείται και υπό την προϋπόθεση ότι το νέο μέλος ε, δήλωσε γραπτά ότι δεν κατέχει άλλη θέση που να αντιβαίνει, να μη συμβαδίζει με την θέση της Ευρωβουλευτού. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. Και τώρα πάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ε, έχω λοιπόν την εξή κατάσταση μπροστά μου. Αυτή τη στιγμή έχουν ζητήσει το λόγο 15 συνάδελφοι. Ε, βεβαίως ε, δεν μπορούμε να δώσουμε το λόγο σε όλους ε, και παρακαλώ να δείξετε κατανόηση γι' αυτό. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ξεκινήσω με τις πολιτικές ομάδες και η πρώτη που θα λάβει το λόγο είναι η κυρία Τσετσεσλεύσκα Γιωχάννα αλλά δεν είναι εδώ στην αίθουσα. Α, εδώ είναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών σε όλη την Ένωση. Ιδίω τώρα που έχουμε την συγκυρία της κρίσης είναι πάρα πολύ σημαντικέ και πρέπει να προσέξουμε και κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ λογικό τώρα να προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε τις αγορές. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο εάν είμαστε συντονισμένοι στα δημοσιονομικά μας. Και θα πρέπει να προσπαθούμε να ρίξουμε το βάρος στην καινοτομία να δημιουργήσουμε θέσει επασχόληση ιδίω για του νέου. να συγκρατήσουμε τι δαπάνε, να αναθεωρήσουμε τις φορολογικές πολιτικές μας και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Και όλα αυτά είναι αποτελέσματα στρατηγικής και προτεραιοτήτων ε, για την Ευρώπη του 2020 και όλα αυτά να τα συντονίσουμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βρούμε διέξοδο σε αυτή την κρίση και πώς θα μπορέσουμε με θετικό τρόπο να βοηθήσουμε την ε, οικονομία μακρόπνο. Η κυρία Μπλινκεπετσούτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών να σκεφτεί τις συνέπειες από την κρίση για την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό που έχουν επιδεινώσει την κατάσταση κάποιων κάτων μελών. Κάποιοι ήδη εφαρμόζουν μέτρα ε, λιτότητας και μάλιστα με ιδιαίτερη επιμέλεια και αυτό έχει πλήξει τελικά τους συνταξιούχους, αυτούς που έχουν μείνει για πολύ καιρό άνεργοι, τους νέους ανέργους. Η φτώχεια των πολιτών σε αυτές τις ε, συνθήκες διαβίωσης όλο και αυξάνεται. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναζητήσουμε θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να τονίσουμε στο Συμβούλιο ότι η διαχείριση του προπολογισμού, τα μέτρα οικονομικής ανάπτυξης, τα μέτρα λιτότητας μάλλον, θα πρέπει να ε, αντισταθμίζονται από μέτρα κοινωνική ανάπτυξης. Διότι όλα αυτά είναι ένα σύνολο και είναι απαραίτητη προπόθεση για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε οι προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού ε, Εξαμήνου, το πακέτο με τα δημοσιονομικά μέτρα και η οικονομική διακυβέρνηση ενισχύουν ουσιαστικά τα μέτρα λιτότητα ε, και εξοφλογισμού που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Η συνταγή αυτή δεν μπορεί να ταιριάζει με τι αρχέ κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη και καταπολέμηση τη ανεργία. Διότι ουσιαστικά μα καταδεικνύουν την αντίθετη κατεύθυνση να εκμεταλλευόμαστε τους εργαζομένους και το κράτος να επιτίθεται στα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, τα οποία ήδη είναι κεκτημένα. Οι πολιτικές λοιπόν αυτές της ε, εδραίωσης των της δημοσιονομικής στήριξης μάλλον, ε, ουσιαστικά λειτουργούν κατά της κοινωνίας και μειώνουν και τα έσοδα των κρατών, τα οικονομικά έσοδα. Θα πρέπει λοιπόν να διακόψουμε αυτή την πορεία. Θα πρέπει συνεργασία μας να έχει κυρίως ε, σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των λαών και την, τον ενεχετισμό των μεγάλων δυνάμεων που πήραν να εκμεταλλεύονται. Στην Πορτογαλία το Σαββατοκύριακο 300.000 ε, άτομα διαδήλωσαν για να σταματήσουν τα μέτρα λιτότητας και πιστεύω ότι η διαμαρτυρία αυτή θα συνεχιστεί. Τσάπα Τσάπα η έκθεση για την ανάπτυξη το 2012 ε, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που ελέγχθηκε και προηγουμένως. Δηλαδή όσον αφορά την ε, κρίση χρέους ε, και την αντιμετώπιση της δεν πρέπει να ξεχνάμε την κοινωνική πτυχή του θέματος. Η κρίση χρέους είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αλλά κατά την αντιμετώπιση της δεν πρέπει να πληγούν οι έτσι κι αλλιώς φτωχοί. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το βιωτικό επίπεδο πρέπει να βελτιώνεται και όχι να επιδεινώνεται. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας κατά την σύνταξη του προεπολογισμού και δεν πρέπει να θυσιάσουμε την ανάπτυξη αλλά ούτε και την ε, κοινωνική ευθύνη. Νομίζω ότι μετά από κάποια χρονιά δεν πρέπει να στρέφουμε το βλέμμα προ τα πίσω και να λέμε ότι το 2012 ήταν η μεγάλη χρονιά τη κρίση. Η κυρία Φλασίκοβα Μπένοβα. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα πρώτα να σας πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ το έργο που επετέλεσε η κυρία Μπερές με την έκθεσή της διότι εκεί δεν αναφέρεται μόνο σε κάποια αρνητικά περιοριστικά μέτρα λιτότητας αλλά αντιμετωπίζει την ε, κρίση όπως είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Η δε προσέγγιση που είχαμε μέχρι σήμερα δεν νομίζω ότι μας βοηθάει και πάρα πολύ. Ε, θα πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε τους στόχους της στατικής μας για το 2020 και για την απασχόληση θα πρέπει να προβούμε σε επενδύσεις, να έχουμε πιο βιώσιμη αγορά εργασίας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις κοινωνικές έγινε ομάδες που περισσότερο χτυπήθηκαν από την κρίση να βοηθήσουμε με διανεμητικό τρόπο την κοινωνία. Άρα, στήριξε στην αγορά απασχόληση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα λιτότητας για να τίθασεύσουν τα δημοσιονομικά. Στην Ιρλανδία, δεκαετία του 80, Κάναμε κάτι τέτοιο και πετύχαμε την ανάκαμψη εγκαίρως. Τώρα, το θέμα είναι να μπορέσει να επιβιώσει ο κόσμος από τη λιτότητα. Άρα, να υπάρξουν και κάποια κίνητρα στην οικονομία. Χρειάζεται όχι μόνο το μπαστούνι αλλά και το καρότο. υπόσταση της Ελλάδας όσον αφορά το ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο τη κοινότητα, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει για να μπορέσουμε να ξεχάσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα, γιατί νομίζω ότι όλοι θα ωφεληθούμε εάν εκτός από τον μπαστούνι έχουμε καρότο, περισσότερο καρότο. Κομισάριο Άντορ, ayer el comisario Oli Rehn aplaudía una reforma en España. Μεταρρύθμιση λέμε ε, που πρέπει να κάνουμε εμείς στην Ισπανία τόσο ώστε να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ε, νέους που έχουν πληγεί από την ανεργία. Είπαμε ο κοινωνικός χάρτης προστατεύει ε, κατά των αυθαίρετων απολύσεων. είπαμε ότι δεν θέλουμε να εξαθλιώσουμε τους εργαζόμενους και θέλουμε αξιοπρεπή δουλειά για τους νέους μας. Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μπίρκα, αυτό που έχει σημασία είναι να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά τα προβλήματα ανάπτυξης και χρέους ε, σε ορισμένα κράτη. Ε, το να κλείνουν τρύπε, αυτό προφανώς ε, δεν είναι η τελική λύση. Ε, πρέπει να υπάρξουν πολλά περισσότερα, να γίνουν επενδύσεις και αυτό εν είδη βοήθειας για αυτοβοήθεια. Επενδύσεις στην παιδεία, στην έρευνα, στην καινοτομία, να παρασκευτεί βοήθεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα πυροδοτηθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση. Απαραίτητο είναι βέβαια να υπάρχει και έλεγχος από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κατά πόσο τα διατηθέμενα κονδύλια χρησιμοποιούνται δεόντως. Μόνο λοιπόν κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θα κατορθώσουμε και εμείς ε, να αποκτήσουμε τη συνένεση κυρίως εκείνων των κρατών μελών ε, που ε, διαθέτουν μεγάλη οικονομική βοήθεια και μέχρι τώρα είχαν χρηστή οικονομική διαχείριση. Η εμπειρία μέχρι σήμερα έχει καταδείξει ότι καλή είναι η εμπιστοσύνη αλλά και η αλληλέγγυα κοινωνία χρειάζεται τον απαραίτητο έλεγχο. Ο κύριος Βίκτορ Ποστινάρο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλα αυτά ακούγονται πολύ ωραία. Οι εκθέσεις που έχουμε μπροστά μας και οι παρεμβάσεις της Επιτροπής ακούγονται πολύ ευχάριστα. Όμως αντιφάσκουν με τη δραματική πραγματικότητα των κρατών μελών. Εκεί οι άνεργοι δεν λαμβάνουν πλέον κανένα κρατικό επίδομα. Δεν αναφέρονται τις στατιστικά στοιχεία και δεν λαμβάνονται και υπόψη στον κρατικό σχεδιασμό πολιτικών. Η μεταρρύθμιση των συνταξιδοτικών συστημάτων, η ευελιξία της αγοράς εργασίας είναι πολύ ωραία λόγια, ακούγονται υπέροχα και είναι σημαντικά. Όμω και στη Ρουμανία, υπό την επιτήρηση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φέραμε ει πέρα μεταρρυθμίσει που σήμεραν την ε, αποδιάρθρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, του κώδικα εργασία και του εργατικού δικαίου και βεβαίω την διάλυση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου. Οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν πλέον δικαίωμα να λαμβάνουν μέρο στον αποκαλούμενο διάλογο Χρειαζόμαστε λοιπόν να ανακάμψουμε και να εξεύρουμε απαντήσεις. Ιδάλλως η Ρουμανία θα είναι ένα μέρος των στατιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Eurostat για το τι συμβαίνει στην επικρατεία της Ευρώπης. Ο... Δεν θα ήθελε να υπάρχει κανείς άνεργος στην Ρουμανία, όσο φιλελεύθερες ε, απόψεις και αν έχουμε. Κανένα ούτε στο Στρασβούργο ούτε στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και τελευταίο ομιλητή στη διαδικασία Κατσέα, ο κύριο ε, Φαία. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω του ε, εισηγητέ των εκθέσεων που συζητούμε, ειδικώ τον συνάδελφο Γκοζέ διότι η έκθεση του υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθούν λύσεις για την οικονομική κρίση, για την δημοσιονομική κρίση που ζούμε τώρα με πειθαρχία αλλά και με μέτρα ανάπτυξης μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης. Θα πρέπει να ορίσουμε προτεραιότητες, να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Μπορεί κάποια πράγματα ε, ε, που φαίνονται αντιφατικά τελικά να μην είναι η λύση. Χρειάζεται να βρούμε λύσεις για την, μεσοπρό... την ευραχυπρόθεσμη κατάσταση, για να τονώσουμε την πραγματική οικονομία. Να επιληθεί το πρόβλημα του τραπεζικού συστήματο που ζούμε αυτή τη στιγμή. Να επιλύσουμε το πρόβλημα των κρατών μελών. Αλλά σε μια δεύτερη φάση θα πρέπει ταυτόχρονα να προβλέψουμε διαρθρωτικέ αλλαγέ, οι οποίε να είναι σαφεί. Σαφεί και να οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη. Τέλο, νομίζω ότι είναι εξίσου αναγκαίο να υπάρξει ένα σύνορο θεσμικών αλλαγών ω προ τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τέλο, χρειάζεται να γίνει σαφή πολιτική συζήτηση. Ποιο στόχο θέλουμε να στηρίξουμε. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και το Συμβούλιο για την παρέμβαση του σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δυστυχώ είμαι τώρα αναγκασμένο να διακόψω αυτή τη διαδικασία Catch the Eye, διότι πρέπει να ακούσουμε και την Κομισιόν, το Συμβούλιο και του συζητητέ. Και στι 12.30 Θέλουμε να ε, ψηφίσουμε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ο κύριος ε, Λάσλο. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να ακούσω τις απόψεις σας για την εκθέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχήν θεωρώ ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων για τις βασικές προτεραιότητες για το 2012. Το ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, η έλλειψη πρωτοβουλειών, όχι απλά να μιλάμε γενικά για την απασχόληση. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερη ε, σχέση, συνδυασμός ανάμεσα σε μακροχρόνια προγράμματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Στατική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βραχυπρόθεσμα. Αυτή λοιπόν η σύγκληση βραχυχρόνου και μακροχρόνων προγραμμάτων είναι πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τους ε, ερετούς ε, εκπροσώπους γιατί έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε καλύτερα μεταρρυθμίσεις και να ε, ενισχύσουμε περισσότερο την εμπιστοσύνη. Ακούστηκαν βέβαια διάφορες πολιτικές απόψεις, προσεγγίσεις και διαπιστώνω ότι και ο καθένας βλέπει διαφορετικά το θέμα των εργαλείων. Υπάρχει μια μεγάλη διάσταση απόψεων. Σίγουρα στόχος ε, είναι η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα μου επιτρέψεις να αναφέρω την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δούμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει για την ανάπτυξη και κυρίως για να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης για την περίοδο, στην περίοδο κατά για την οποία μιλάμε. Κατά τη συζήτηση ε, φάνηκε ότι ε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερες ευκαιρίες ε, και είμαι ευγνώμων για τις θετικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της Επιτροπής. Εμείς ξεκινήσαμε μία προεκλογική εκστρατεία για την προσφορά εγκυρίσεων, εγγύσεων στους νέους. Ε, Έρη Πάστος Κούρμα, ευχαριστώ πολύ ε, που ανέφεραν αυτή την εγγύηση και τη σχολήσαν με θετικά λόγια. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παράσχει τεχνική βοήθεια στα κράτη-μέλη τα οποία είναι πρόθυμα να ακολουθήσουν αυτό τον δρόμο. Επίσης, ε, όπως ανέφεραν και πολλοί άλλοι μετέχοντες στη συζήτηση, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η παιδεία και η κατάρτιση, καλύτερη ταύτιση να υπάρχει ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά εργασία. Και αυτό θα καλυφθεί στι ειδικέ συστάσεις των κρατών μελών ε, στο τέλος ε, του εξαμήνου. Όμως, επειδή ε, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία των νέων, ε, εργαζόμεθα και για την ε, ε, επικαιροποίηση της πολιτικής απασχόλησης έτσι ώστε τον Απρίλη να κατατεθεί ένα πακέτο απασχόλησης το οποίο θα ανταποκρίνεται σε πολλά θέματα που δείξατε πώς οι πολιτικές παρήματος χάρη της ευελιξίας και της ασφάλειας επηρέασαν την αγορά εργασίας εμπνευστήκαμε από την Δανία αλλά θέλουμε και να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε περισσότερο και αποτελεσματικότερα για να δημιουργηθούν πράσινες θέσεις απασχόλησης. Αυτός είναι ένας από τους ε, τομείς ε, που θα ενισχυθεί περισσότερο στο μέλλον. Θα ενισχύσουμε ε, την πράσινη απασχόληση στην Ευρώπη και σε άλλες υπήρους, γιατί αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Πέρα από τις πράσινες θέσεις απασχόλησης, πρέπει να δούμε και άλλες θέσεις απασχόλησης, κυρίως στον τομέα της πληροφορικής. Η πληροφορική θα είναι μεγάλος εργοδότης στο μέλλον. Αυτό λοιπόν το πακέτο αυτό περιλαμβάνει πάρα πολλές ε, πρωτοβουλίες. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και αποτελεσματικότερα για ποιοτικέ ε, θέσεις εργασίας και για την προσφορά ευκαιριών στους νέους. Αυτό το ποιοτικό πλαίσιο θα αποτελέσει εργαλείο κλειδί ε, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Είναι λοιπόν απαραίτητα να γίνουν περισσότερα για τις επιχειρήσεις, κυρίως για τις ε, μικρομεσαίες. Σημαντικό αυτό. Ας δούμε όμως ποιο είναι το πραγματικό αδιέξοδο όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τις ε, μικρομεσαίες. Ίσως μπορεί κανείς να θεσπίσει καλύτερη ε, καλύτερους κανονισμούς, αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο τραπεζικός τομέας θα χρηματοδοτεί καλύτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικότερα επιχειρήσεις. Να προσφέρουμε μικροοικονομικές δυνατότητες αυτό πρέπει να εισαχθεί ε, σε πάνω από ένα τρίτο των κρατών μελών και εργαζόμαστε και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη πέραν του ενό τρίτου για να ε, εισαχθούν μικροχρηματοδοτικέ δυνατότητε στο συντομότερο δυνατόν. Επίση, επιτρέψτε μου να πω ότι κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πρόκληση στην οικονομική διακυβέρνηση είναι η αυξανόμενη πόλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται μόνο για διαφοροποίηση. Ε, εφαρμόζουμε την αρχή ότι δεν μπορεί ένα πράγμα να ταιριάζει για όλου. Ε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα τη διαφορετικότητα. Όμω τώρα βιώνουμε κάτι που είναι πολύ πιο σοβαρό. Βλέπουμε μεγαλύτερη ασυμμετρία, πόλωση ανάμεσα στα κράτη-μέλη που είναι ισχυρά, ε, με απασχόληση και κοινωνική σταθερότητα, αυτή από τη μια και από την άλλη τα κράτη-μέλη τη ε, περιφέρεια, όπου όλα αυτά είναι πολύ πιο δύσκολα και αντί για ανάκαμψη, δυστυχώ πολλά κράτη-μέλη βιώνουν για εφέτο ύφεση ε, και υπάρχει κίνδυνος να χαθεί μία γενιά. Για πολλά κράτη-μέλη, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, υπάρχει μάλιστα ε, και σημαντική ροή μετανάστευσης. Φεύγουν οι νέοι από την Ευρώπη γιατί δεν βλέπουν να υπάρχουν για αυτούς ευκαιρίες και δεν θεωρούν ότι θα επανέλθουν τα επόμενα χρόνια. Είμαι επίσης ευγνώμων και για το σχόλιο που έγινε από τη Λετωνία γιατί φάνηκε ότι παρότι επανήλθε κάποια σταθερότητα δεν θα πρέπει αυτό το παράδειγμα να χρησιμοποιείται ως ε, μοντέλο για άλλες χώρες που αναζητούν την έξοδο από την ύφεση και την επίτευξη χρηματοψητικής σταθερότητας. Κυρίες και κύριοι, θέλω να υπογραμμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι μια διαδικασία μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους. Ε, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, πήραμε σημαντικά μαθήματα, διδαχτήκαμε πολλά και βεβαίως διαπιστώσαμε ότι υπάρχει και μεγαλύτερο περιθώριο για συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ανοιχτή συζήτηση και δημοκρατική ε, λογοδοσία για να επιτύχει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τη στρατηγική τη ε, οικονομικής διακυβέρνησης. θέλουμε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των στόχων απασχόλησης ε, και των κοινωνικών στόχων, να εφαρμοστεί μια τέτοια πολιτική που θα οδηγήσει στην επιτυχία. Όλα αυτά αφορούν ε, στην στρατηγική Ευρωπαϊκή Ευρώπη 2020, αφορούν το περιεχόμενό της, τους αριθμούς. Δεν πρέπει να τα εγκαταλείψουμε όλα αυτά. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε και εσάς ε, να μας βοηθήσετε να ενισχύσουμε τη σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια έτσι ώστε τους στόχους του 2020 να τους μεταφέρουμε και να τους συμπεριλάβουμε και στις εθνικές στρατηγικές. Ευχαριστούμε, ο Πρόεδρος, ε, ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε, για την απάντησή σας και τώρα έχει το λόγο κυρία Βεσταγέτσε εκ μέρους του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν με ρωτήσουν οι κόσμοι του τύπου φεύγοντα από αυτή την αίθουσα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα τη συζήτηση και ποιο το νόημα, θα έλεγα η ανεργία των νέων. Νομίζω αυτό ήταν ε, το καθοριστικό για τον κάθε από τον ομιλητή. Για όλε αυτέ τι ώρε που συζητήσαμε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Νομίζω ότι είναι καθοριστικό σημείο και θα πρέπει να βρούμε έναν αποτελεσματικό τρόπο να επιλύσουμε το θέμα αυτό φαίνεται ότι δεν υπάρχει απαραίτητο αντίφαση μεταξύ της ε, εδραίωση τη δημοσιονομική και τη ανάπτυξη. Το θέμα είναι τι θα τεθεί ω προτεραιότητα. Είναι δύσκολο, δεν θα είναι απλό να βρούμε λύση, αλλά θα πρέπει να τεθούν σωστά προτεραιότητε. Διότι το θέμα δεν είναι απλώς πώ θα ξοδέψουμε το επόμενο και το επόμενο δισεκατομμύριο, αλλά πώ θα το ξοδέψουμε ευφυώ, ώστε να γίνουν δαπάνε κατά τρόπο σωστό. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και για το Ευρωκοινοβούλιο και για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι σωστέ οι προτεραιότητέ μα. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Η ερώτηση ουσία. Και νομίζω ότι εκεί θα υπάρξουν πολλέ διαφωνίε. Διότι αν θέλουμε να αλλάξουμε τι προτεραιότητέ μα, θα πρέπει να αλλάξουμε κάποιο από τα συστατικά που αλλάζουν βεβαίω και το ποιοι είναι οι σημερινοί δικαιούχοι των σημερινών δαπανών των των προπολογισμών. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι μέρο τη λύση είναι να γίνει πιο οικολογική η οικονομία μα. Κάποιοι λένε να περιμένουμε. Όχι. Το να γίνει πιο οικολογική η οικονομία μα είναι μέρο τη απάντηση. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο πώ χρησιμοποιούμε του πόρου μα. Και για τον σκοπό αυτό θα δημιουργήσουμε και περισσότερο χώρο για, την βασικότερη, για το βασικότερο από τους πόρους μας, τα ανθρώπινα όντα, τους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν οι πέντε προτεραιότητε που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τεθούν σε σωστή σειρά. Οι πέντε προτεραιότητε επιτροπής είναι καθοριστικά βήματα για να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής της Ευρώπης το 2020. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι επιδιώκουμε διαφοροποιημένες ε, διαφοροποιημένα μέτρα με σκοπό την φορολογική ανάλυση που να επιτρέπουν και την ανάπτυξη. Επίση, καμία μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να δημιουργήσει θέσει εργασία εάν δεν μπορεί να δανειστεί, εάν κοπεί η πιστοτική τη γραμμή. Είναι λοιπόν σημαντικό και να υπάρχουν μέτρα δανεισμού και να επιτρέπουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και για το μέλλον. Νομίζω πολλές προτάσεις έχουν ήδη υποβληθεί που υποδεικνύουν ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Τέταρτον, και επειδή το συζητήσαμε διαμακρόν σήμερα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και τι κοινωνικέ επιπτώσει τη κρίση. Και πέμπτον, ίσω κάτι που έχουμε υποτιμήσει ελαφρώ, ο εξυγχρονισμό των κρατικών μηχανισμών. Θα πρέπει να επιτρέπουμε και στις επιχειρήσεις να δημιουργούν θέσεις εργασία. Νομίζω αυτά είναι τα σημεία ουσία και νομίζω η αγορά εργασία θα πρέπει να μελετηθεί ώστε να καταλάβουμε πώ θα διευκολύνουμε την είσοδο των νέων στην αγορά εργασία. Θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στι επιχειρήσει και να μπορούν να συμμετέχουν. Να καταλαβαίνουν ότι η δουλειά τους ωφελεί και τις ίδιε τι επιχειρήσεις σε αντάλλαγμα. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, νομίζω η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι θα ξαναγίνει επανειλημμένο στο μέλλον. όπως έχει γίνει και στο παρελθόν η περίοδος της κρίσης και η αντιμετώπιση της είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και είναι επώδυνη για όλους. Αλλά χρειάζεται εδώ συντονισμό. Και όταν συζητούμε τις λύσεις πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποια από τα πράγματα που ανέφερα εγώ και από αυτά που ανέφερε ο Επίτροπος και από τα στοιχεία των παρεμβάσεων σήμερα. Η πραγματική πρόκληση είναι να βεβαιωθούμε ότι θα συνεργαστούμε πραγματικά. Ανυπομονώ να συνεχίσω την σχέση συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο, να λάβω υπόψη τι προτάσει που ήδη έχουν υποβληθεί και να επωφεληθούμε από όσα αναφέρονται. Δεν υπάρχει αναγκαστικά αντίφαση μεταξύ τη συνετή ευρέωση και τη ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, τελειώνει λοιπόν η συζήτηση με τους ε, εισηγητές και οι πρώτη που έχει ζητήσει το λόγο είναι η κυρία Κορνέλισεν. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους σας για αυτή τη συζήτηση. Και τους και οι οποίοι συνεργάστηκαν ε, με τρόπο θετικό και διεκπαιρεωτικό, Γκοζές και Μπερές, επίσης άλλοι που πρέπει να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία τους, ε, για εκείνους κάναμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη τρόικα, ένα τρίο πάρα πολύ πετυχημένο επίσης. Έτσι μπορέσαμε να αλληλοσυμπληρώσουμε τις απόψεις για το οικονομικό τοπίο και επίσης ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που γενικότερα τώρα στην Ολομέλεια να στηρίξατε κύριε Χάουγκ επίσης θα πρέπει να καλύψουν όλες τις χώρες και τις χώρες που έχουν το, το, το έλλειμμα και το χρέος ε, επίσης οι πλεονασματικές χώρες ε, ε, και αυτές θα πρέπει να καλυφθούν όπως η Ολλανδία και η Γερμανία και είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση ασύμμετρου χαρακτήρα. Επίση, θα πρέπει να δούμε πώ θα ανακτήσουμε τι χαμένε θέσει εργασία, να αντιμετωπίσουμε επίση την φτώχεια, κάτι το οποίο το έχουν υπόψη του όλε τι μικροοργανώσει, πολιτικέ ομάδε θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα, μένουμε μόνο στα λόγια όπως μέχρι σήμερα. Μέτρα για κοινωνική πολιτική και έτσι να μπορέσουμε με τα απαραίτητα συνοδευτικά μέτρα να πλαισιώσουμε τα δημοσιονομικού χαρακτήρα μέτρα. Εκτός από την εξαπλή δεσμή μέτρων θα πρέπει να έχουμε τι, οκταπλή, δεκαπλή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Με διαφοροποιημένη στρατηγική, επομένως, να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα κατημέρια και να τα οδηγήσουμε στην ανάκαμψη της οικονομίας. Γκοζές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω και τώρα δεν είναι η καλύτερη στιγμή να λαμβάνει κανεί το λόγο, αλλά θέλω και εγώ να σα πω ότι ήταν πάρα πολύ αγαστή η συνεργασία μεταξύ τη κυρία Κορνέλη, τη κυρία Μπερέ και του ομιλούντο. Επί τη ουσία, θα πρέπει να σα πω ότι αυτό που σήμερα χρειαζόμαστε είναι να συνοδεύσουμε του λόγου με τα έργα. Και βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο τώρα, ε, διαδικαστικό, τυπικό. Η χρήση του 2012 ε, θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε αυτό το νέο ε, αριθμιστικό πλαίσιο της ενισχυμένης ε, οικονομικής διακυβέρνησης. Οπότε θέλω κύριε Επίτροπε να σας πω ότι χρειαζόμαστε από πλευρά σας μια έκθεση εντελεχή όσον αφορά ε, της, ε, το τι, ισχύει για κάθε χώρα και το Συμβούλιο θα πρέπει δημοσία να διατυπώσει τη θέση του όσον αφορά τον οικονομικό διάλογο με το Κοινοβούλιο, διότι αφίστανται οι θέσεις μας σε σχέση με τις προτάσεις της Κομισιόν. Και βεβαίως τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο ελιγμών ε, και πρέπει να απολάβουν τις ε, επικουρικότητες. Το νέο αυτονομικό πλαίσιο προβλέπει ότι θα πρέπει να εμπλέκεται σημαντικά σε αυτό το ε, ευρωπαϊκό εξάμεινο το κοινοβούλιο με διαφάνεια, με υπευθυνότητα να λαμβάνονται έτσι οι αποφάσεις και κυρίως όσον αφορά τον οικονομικό διάλογο όπως ε, όπως ορίζεται και όποτε χρειάζεται. Επίσης θα πρέπει να σας υπενθυμίσω αυτά τα οποία έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο επισήμως προς Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εκείνο το ψήφισμα της 1ης 12 του 2011 και θα πρέπει επομένω να δοθεί απάντηση σε αυτό που ζητήσαμε εκείνο το ψήφισμα με τρόπο συγκεκριμένο ρεαλιστικά και αποτελεσματικά να ασκείται ο δημοκρατικός έλεγχος που δικαιούται να ασκεί αυτό εδώ το Κοινοβούλιο. Τελείωσε λοιπόν η συζήτηση ή τελειώνει με την εισηγήτρια κυρία Περές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μας είπατε ότι το Ευρωκοινοβούλιο δέχτηκε να μην αλλάξουν οι κατευθυντήριες γραμμές. Έστω όμως θα θέλαμε οι κατευθυντήριες γραμμές επιτέλους να υλοποιηθούν στην έκθεσή μας κάνουμε μια σειρά από προτάσεις ώστε να έχετε κι εσείς τρόπο να επιβλέπετε αυτήν την υλοποίηση. Κυρίως θέλω να σταθώ σε μία από τις προτάσεις. Να συνεργαστείτε με τα κράτη-μέλη ώστε να υπάρχει ονοματολογία δημοσιονομική που να επιτρέπει να διαπιστώνεται η συμβολή των κρατών μελών λόγω χάρη στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής του 2020. Όχι στα ιδιωτικές δαπάνες λόγου χάρη όπως τώρα τις γνωρίζουμε. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την ε, προθυμία σας και τον τρόπο που μας είπατε ότι στο ΕΚΟΦΗΝ ε, της 21ης Φεβρουαρίου θα λυθεί υπόψη η συζήτηση αυτή και το έργο του Κοινοβουλίου. Αυτό ακριβώς επιθυμούμε. Ακριβώς αυτό είναι το πνεύμα μας και έτσι θέλουμε να προχωρήσει η δημοκρατία στην Ευρώπη. Ακριβώς σε αυτό το το οποίο θέλουμε στις 27 και 28 Φεβρουαρίου να συναντήσουμε τους εκπροσώπους όλων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Διότι στο ευρωπαϊκό αυτό εξάμεινο θέλουμε δημοκρατική διάσταση επιτέλους να λάβει σάρκα και ουστά. Κυρία Υπουργέ, επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου να σας απευθύνω μία έκκληση. Κατά το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ κατά τον ίδιο τρόπο να λάβετε υπόψη τη νέα μελέτη αντικτύπου που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει λογικά αύριο προκειμένου να αξιολογήσει την δυνατότητα φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρίες και κύριοι. Τελειώνει λοιπόν η κοινή συζήτηση για το θέμα ε, ανάπτυξης και απασχόλησης. Παρακαλώ λοιπόν να καθίσετε όλοι για να ξεκινήσουμε αμέσως με την ψηφοφορία.